ότι υπάρχει μια προσπάθεια παραβίαση των δικαιωμάτων των γυναικών. Το, κοινοβου... το Συμβούλιο θα πρέπει να πάρει θέση και να επιλέξει. Θα ήθελα, ε, συγγνώμη, θα ήθελα να ζητήσω ε, από τα μέλη να τηρήσουν το χρόνο ομιλίας. Η επόμενη ομιλήτρια είναι η κυρία Λουκατσέσκα. Ευχαριστώ πολύ. η έκθεση εργασίας του Oxfam η έκθεση των, του Oxfam συγγνώμη, είναι πολύ ξεκάθαρη όσον αφορά την, ε, την εκμετάλλευση των γυναικών. Οι γυναίκες είναι αυτές που κάνουν τα τρία τέταρτα μη πληρωμένης, μη αμοιβόμενης ε, εργασίας ε, στο σπίτι και με τα παιδιά η ίση αμοιβή αφορά και τις γυναίκες με αναπηρίες, ηλικιωμένες γυναίκες, ε, η συρρήκνωση ε, του αριθμού των γυναικών στην αγορά εργασίας ε, διαπιστώνεται παντού. Η επιδείνωση της κλιματικής αλλαγής στην κατάσταση των γυναικών και αυτό είναι ένα θέμα μεταξύ όλων όσων προανέφερα που θα έπρεπε να συζητηθούν στο επίπεδο των Ηνωμένων Εθνών προκειμένου να αναλυφθούν πολιτικές δεσμεύσεις. Η κυρία Μάρκες, για ένα λεπτό. Η ισότητα είναι θέμα εξουσίας. Η εξουσία δεν δίνεται. Πάντα πρέπει να την κατακτήσεις. Δεν θέλουμε να συνδυάσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα με την ισότητα των γυναικών ε, προ όφελο των γυναικών. Αυτό είναι προ όφελο και των ανδρών και των γυναικών. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ μιλάει για έναν άντρα ο οποίος ήταν πάντα φεμινιστής. Ποιες είναι οι προτεραιότητες του ΟΗΕ 25 χρόνια μετά το Πεκίνο. Καταρχάς, τον αγώνα υπέρ των γυναικών που δεν έχουν δικαίωμα. Δεν έχουν δικαίωμα να σπουδάσουν, να παντρευτούν. Δεν έχουν δικαίωμα να ελέγξουν τη σεξουαλική του ζωή. Που δεν έχουν δικαίωμα να έχουν επαγγελματική ζωή. Αυτέ τι γυναίκε θα πρέπει να τι κάνουμε προτεραιότητά μα. Εν συνεχεία, προτεραιότητα είναι να καταπολεμήσουμε τη βία. Ε, επίσης και τη νέα μορφή βίας που υπάρχει στο ίντερνετ που αγγίζει πάνω απ' όλα τις γυναίκες και τα κορίτσια. Επίσης, υπάρχουν και άλλες ανισότητες. Αυτές που είναι σήμερα ανισότητες και, σήμερα, και θα συνεχίσουν να είναι ανισότητες αν υπάρχει πρόληψη. Όπως παραδείγματο χάρη ε, η ανισορροπία της παρουσίας ανδρών και γυναικών στα τεχνολογικά επαγγέλματα. Έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε σε όλο τον κόσμο και αν είμαστε ενωμένοι θα είμαστε πιο δυνατοί. Ευχαριστώ. Ζητάμε ακόμα μια φορά να σεβαστείτε το χρόνο μιλία σας. Η κυρία Ζαχαροπούλου 1,5 λεπτό. Κυρία Επίτροπε, κυρία Υπουργέ, όπως ξέρετε, τα δικαιώματα της σεξουαλικής υγείας και της αναπαραγωγικής υγείας είναι σημαντικό θέμα για να υπάρξει ισότητα άνδρων και γυναικών. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μία υπαναχώρηση σε πολλά σημεία του πλανήτη και συχνά με την υποστήριξη μεγάλων κρατών όπως οι ΗΠΑ, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση χάνει, αυτή την αξιοπιστία τη αν δεν μιλήσει για αυτά τα θέματα με μία κενή φωνή. Παραδείγματο χάρη σύνοδο κορυφής του Ναϊρόμπι τον Νοέμβριο για τη διάσκεψη του ΟΗΕ για το, τους πληθυσμούς και την ανάπτυξη. Εγώ βρήκα σοκαριστικό και απαράδεκτο το ότι η Πολωνία και η Ουγγαρία, δύο κράτη-μέλη, συντάχθηκαν με εκείνου που αμφισβητούν τα δικαιώματα των γυναικών. Κυρία Επίτροπε, κυρία Υπουργέ, οι νέε γενιέ δεν ήταν ποτέ τόσο συνειδητοποιημένε για το θέμα της ισότητας ανδρών και γυναικών. Ε, και σε όλο τον πλανήτη φωνάζουν στη Χιλή, στο, στην Αργεντινή, στο Μεξικό, στην Ισπανία, στη Γαλλία, στο Βέλγιο. Παντού στον κόσμο. Γιατί αυτή η γενιά δεν δέχεται πια αυτή την ε, αδικία. Αυτή είναι η γενιά της ισότητας. Και ενώ γιορτάζουμε την 25η ε, χρονιά από τη δήλωση του Πεκίνου, θα πρέπει μαζί με αυτούς τους άντρες και τις γυναίκες, με αυτά τα κορίτσια και τα γόρια που απο, αποαπητούν μια δίκαιη κοινωνία, μια ίση κοινωνία, να συνταχτούμε και εμείς με αυτούς. Αυτή είναι η Ευρώπη, αυτέ είναι αυτές είναι οι αξίες μας και αυτό πρέπει εμείς ως πολιτικοί να προωθήσουμε. Η κυρία Μπρούνα, για μισή λεπτό. Πρόεδρε, ευχαριστώ πρέπει να καθορίσουμε τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά τις συνθήκες για, τους, για τις γυναίκες. Η αντιπροσωπεία μας θα μιλήσει για ίση αμοιβή, για ίση εργασία, κατά της βία στο ίντερνετ, της, τους αναγκαστικούς γάμους και τον ακροτηριασμό των γυναικό, γεννητικών οργάνων. Θα πρέπει να αναγνωρίσετε η δουλειά που κάνουν οι γυναίκες στο σπίτι και δεν θα ψηφίσουμε το ψήφισμά σας που είναι καρικατούρα ε, δεν θέλουμε να αμφισβητηθεί η σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Ε, ένα βασικό θέμα ε, είναι για σας ταμπού. Το βάρος του ριζοσπαστικού Ισλάμ παντού σε όλο τον κόσμο. Στη Γαλλία η Μίλα ε, ένα κορίτσι, επειδή κριτήκανε το Ισλάμ, δέχτηκε επίθεση στο λύκειό της. Έλαβε ε, εκατοντάδες ε, απειλές θανάτου, επιθετικά μηνύματα και δεν μπόρεσε να ξαναπάει στο σχολείο, γιατί δεν ήταν ασφαλής. Και την φυλάει η αστυνομία τώρα. Μετά από τρεις εβδομάδε που δεν πάει στο σχολείο, άλλαξε σχολείο. Αυτή, αυτό το κορίτσι είναι η καθημερινότητα διαφόρων γυναικών που υφίστανται την επιρροή του ριζοσπαστικού Ισλάμ. Οι φεμινιστέ δεν είπαν τίποτα για αυτό το θέμα. Ταμπού προφανώ για αυτού. Εμεί ζητάμε μια συζήτηση σε αυτή την ολομέλεια και μα αρνήθηκαν να κάνουμε αυτή την ε, συζήτηση. Αλλά πρέπει να ανοίξετε τα μάτια σα για την ε, ε, μετανάστευση και για το ριζοσπαστικό Ισλάμ και πώ επηρεάζει τη ζωή στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Κυρία Ρίβα Ιχινέρ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πίτροπε, κύριε Υπουργέ. Ε, ζούμε σε μια εποχή όπου πολλά δικαιώματα τα οποία θεωρούμε ότι είναι κατοχυρωμένα τελικά αμφισβητούνται. Μια ε, εποχή όπου υπάρχουν ε, ξενόφοβες ε, τάσεις που προσπαθούν ε, να παρεμποδίσουν ε, την πρόοδο προς μια πιο δίκαιη κοινωνία. Και αυτό επηρεάζει αρνητικά ιδιαίτερως εμάς την, ε, τις γυναίκες. Η 64η επέτειος είναι... Ε, η 64η συγγνώμη, Σύνοδος της Επιτροπής του ΟΗΕ είναι μια θαυμάσια ευκαιρία ε, προκειμένου να επιτευχθεί ε, μια πρόοδος πολλοί στόχοι που έχει καταρτήσει η πλατφόρμα για τις ε, γυναίκες είναι σημαντικές γιατί η Ευρώπη θα πρέπει να φρενάρει την ε, παγκόσμια οπισθοδρόμηση όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών. Η επικύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης και η έγκριση του, ε, του συστήματος των ποσοστώσεων ε, ακόμα έχουν τελματώσει στους κόλπους του Συμβουλίου. Θα πρέπει να ασκήσουμε πίεση για να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Η κυρία Μαζούρεκ, για ένα λεπτό παρακαλώ. Κυρίε, Κυρίες, ευχαριστώ πολύ. Πέρασαν 25 χρόνια μετά την Παγκόσμια Σύνοδο του Πεκίνου. Η συζήτηση δείχνει όμως ότι πολλά πρέπει να γίνουν ακόμα για να προστατεύσουμε τις γυναίκες σε πολλές περιοχές. Πρέπει να απαντήσουμε τι έχουμε πετύχει μέχρι τώρα και τι πρέπει να γίνει ούτως ώστε όλες οι γυναίκες να μην αντιμετωπίζουν προβλήματα όπως βία, οικονομική ανισότητα, διακρίσεις των ε, γυναικών ως μητέρες στην αγορά εργασίας. Ίσως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να ακολουθήσει το πολωνικό παράδειγμα όπου ε, το μισθολογικό χάσμα είναι το μικρότερο στην Ευρώπη και η βία ε, δείχνει ότι η Πολωνία είναι από τις ασφαλέστερες χώρες στην Ευρώπη. Είμαστε κατά των ε, αμβλώσεων ως μέτρο οικογενειακού προγραμματισμού και δεν θέλουμε η Ευρώπη να χρηματοδοτεί οργανώσεις που θέλουν την άμβλωση. Τι προτιθέμεθα να κάνουμε στο Κοινοβούλιο όμως για να προστατέψουμε καλά τα δικαιώματα των γυναικών και να έχουμε ισότητα των φίλων. Περιμένω το χρονοδιάγραμμα και την ενημέρωσή σας για τα σχέδια στο μέλλον. Η κυρία Φράνσεν, ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι. Η ισότητα των φύλων δεν είναι κάτι που σταματά στα σύνορα της Ένωσης. 24 χρόνια μετά το Πεκίνο, 25 χρόνια μετά, ε, οι γυναίκες ε, δίνουν μάχη για τη θέση που τους αξίζει. Ε, θέλουμε ε, εκπροσώπησης διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Θέλουμε ε, ισότητα σε όλους τους τομείς. Η επόμενη σύνοδος στη Νέα Υόρκη μας επιτρέπει να αναδείξουμε την θέση των ευάλωτων γυναικών που απειλούνται, που είναι φτωχές, που είναι σε εμπόλεμες ε, περιοχές που πέφτουν θύμα εκμετάλλευσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να μιλήσει με ενιαία φωνή εδώ και μάλιστα με στεναρή φωνή. Ε, πέρασα από την πόρτα της ευκαιρίας ε, και ε, δίνω τις, θέλω να δώσω τις ίδιες ευκαιρίες σε άλλες γυναίκες για να πετύχουν. Και κυρία Μωρέτη, ένα λεπτό. Πέρασαν 25 χρόνια από τη δήλωση του Πεκίνου. Αλλά οι διακρίσεις λόγω φύλου δυστυχώς συνεχίζονται. Ακόμα και σήμερα όταν βιάζεται μια γυναίκα, συζητάμε το πώς δινότανε. Μερικές ε, γυναίκες σε κάποια κράτη-μέλη δεν μπορούν να έχουν ε, δικαίωμα στην άμβλωση. Ε, στην Ευρώπη οι γυναίκες κερδίζουν 16% λιγότερο από τους άντρες. Και αυτό θεωρείται φυσιολογικό. Είναι επίσης φυσιολογικό να σταματάει την καρδιά της μια γυναίκα. Επί 25 χρόνια απλώς λέγαμε λόγια και ένα περιεχομένου. Σήμερα, λίγο πριν τη διάσκεψη του ΟΗΕ, θα ήθελα η Ευρώπη με μία φωνή να διατρανώσει ότι δεν δεχόμαστε πια κάτι τέτοιο. Τα δικαιώματα, τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά των γυναικών θα πρέπει να εξασφαλίζονται παντού. Κυρίως η πρόσβαση σε αντισύλληψη, σίγουρη και νόμιμη άμβλωση, υγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση στα σχολεία. Η ισότητα των φύλων θα πρέπει να μπει στο κέντρο της ε, πρόκλησης κλιματικής αλλαγής. Γιατί οι γυναίκες θα τιμωρηθούν περισσότερο. Έχω εμπιστοσύνη σε εσά, Επίτροπε. Είσαστε γυναίκα. Θέλω να δώσετε το προβάδισμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτά τα θέματα. Η κυρία Αντουέλ. Ε, προτιμώ από το μικροστικό σας ε, φεμινισμό, προτιμώ την πραγματικότητα. Τι κάνετε για να σώσετε τη ε, ζωή των γυναικών, ακροτηριασμός των γυναικών, βιασμοί, συνεχείς φρικαλαιότητες κατά των γυναικών. Γιατί μιλάτε στα Ηνωμένα Έθνη. Ε, είπατε ότι το θέμα των βιασμών χρησιμοποιείται από τους λαϊκιστές ή ε, γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευση στο Πακιστάν από τους ρατσιστές. Ε, οι φεμινιστές που καταδικάζουν μια, ε, ένα παιδί, μια, ένα κοριτσάκι το οποίο στην Γαλλία επειδή είναι από το Ισλάμ. Οι γυναίκες είναι για σας μόνο ενδιαφέρουσε στο βαθμό που είναι ψηφοφόροι. Θα πρέπει να βρείτε το κουράγιο να δείτε ποια είναι η θέση των γυναικών στην ιστορία. Mrs. Klotz, one minute. Your, mic your microphone is not on. Klotz, δεν έχετε μικρόφωνο αναμένο. Ε, Πρόεδρε, στην προφορική ερώτησή τη, η κυρία Ρέγνερ είπε ότι 25 χρόνια μετά τη δήλωση του Πεκίνου ε, τα δικαιώματα των γυναικών δεν γίνονται πλέον σεβαστά. Και εγώ συμφωνώ με αυτό. Γιατί υπάρχουν φο... ε, γυναίκες χωρίς φωνή, χωρίς φωνή και δεν μπορούν να αποφασίσουν για το μέλλον του. Υπάρχουν ε, γυναίκε που η επιβίωσή του. ε, αποφασίζεται από τι μητέρε του, οι οποίε λαμβάνουν υπόψη μόνο τη δική του κοινωνική και οικονομική κατάσταση. Επίση, υπάρχουν ε, γυναίκε που τα σώματά του ε, ακροτηριάζονται χημικά ή φυσικά και σκοτώνονται χωρί καμία συνέπεια για του δράστε. Αισθάνεστε εξοργισμένοι? Θα έπρεπε. Γιατί εκατομμύρια αγέννητα κορίτσια δεν έχουν το δικαίωμα να πολεμήσουν, ε, δεν μπορούν να διαλέξουν το μέλλον τους. Ε, και όμως θα πρέπει να το διαλέξουν, να μπορούν να το διαλέξουν το μέλλον τους. Κανένας ε, άνθρωπος δεν θα πρέπει να στερείται το δικαίωμα να διαθέσει το θέμα του όπως θέλει. Ε, οι κινήσεις, ε, τα κινήματα τα οποία υποστηρίζουν μόνο την ε, άμβλωση και δεν υποστηρίζουν τις γυναίκες, νομίζω ότι είναι βαρβαρικά. Η κυρία σχετικά είναι ένα λεπτό. Από τη δήλωση του Πεκίνου, τα δικαιώματα των γυναικών έχουν προχωρήσει, αλλά έχουν υποστεί και οπισθοχώρηση. Δεν μπορούσαμε να σημειώσουμε πρόοδο σε συμβάσεις διεθνώς. Δεν έχουμε περισσότερες γυναίκες στην πολιτική, δεν έχουμε γυναίκες σε ηγετικές θέσεις. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε τις ποσοστώσεις. Ξέρουμε την, τον αγώνα που δίνουν οι οργανώσει των γυναικών ε, για τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα, αλλά η μάχη αυτή έχει αποδυναμωθεί παγκόσμια. Γι' αυτό στρέφομαι με ελπίδα προς την Επιτροπή, γιατί θα πρέπει αυτό το πρόγραμμα για την ισότητα να προχωρήσει. Και ελπίζω να, παίζετε, να παίξετε ηγετικό ρόλο παγκόσμια, ούτω ώστε να βάλετε τα δικαιώματα των γυναικών και τα ανθρώπινα δικαιώματα στις διαπραγματεύσεις. Ε, με βάση τους βιώσιμους στόχους της ανάπτυξης, να κάνετε μελέτη αντικτύπου για τη διάσταση του φύλου σε όλες τις πολιτικές και να λάβετε υπόψη σας την σύμβαση της ε, ε, Κωνσταντινούπολης, να λάβουμε υπόψη μας και την Αφρική και να δώσουμε και καλύτερη χρηματοδότηση σε ΜΚΟ που πολεμούν για τα δικαιώματα των γυναικών. Η κυρία Κονσάλες για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, η δήλωση του Πεκίνου 25 ε, χρόνια μετά είναι ο δείκτης για να προσμετρήσουμε τις ανισότητες του φύλου. Αλλά είμαστε ρεαλιστές. Πολλές χώρες ε, ε, πολλές από αυτές τις αρχές δεν εκπληρώνονται οι συνεδρίες του ΕΕ είναι μια καλή ευκαιρία για να προεπισπιστούμε συγκεκριμένα πράγματα, τα αναπαραγωγικά και σεξουαλικά δικαιώματα των γυναικών, συγκεκριμένα των γυναικών που ζουν στη Λατινική Αμερική, από την προοπτική της ε, εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, πέρα από την ανισότητα, κάτω από οικονομικέ ε, προποθέσει όσον αφορά βασικά δικαιώματα όπω είναι η ζωή, η σωματική ακαιρεότητα, η σεξουαλική ελευθερία και η αναπαραγωγική υγεία. Στην ε, Λατινική Αμερική και στην Καραϊβική υπάρχουν τα υψηλότερα ποσοστά παράνομων αμβλώσεων και θανάτου κατόπιν παράνομων ε, αμβλώσεων. Ε, έξι χώρες ε, απαγορεύουν τις αμβλώσεις και οι αμβλώσεις γίνονται με κέντρο της ζωής των γυναικών. Ε, τα Ηνωμένα Έθνη θα πρέπει να υποστηρίξουν οργανισμούς ε, οι οποίες προσπαθούν να προστατεύσουν τις γυναίκες. Η αντισύλληψη για να μην προχωρήσουν στην άμβλωση ή άμβλωση και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να δούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Η επόμενη αμιλήτρια είναι η κυρία Φερακούτ για ένα λεπτό. Ε, ευχαριστώ. Ε, γιορτάσουμε την 64η Σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ. 25 χρόνια μετά τη δήλωση του Πεκίνου, ε, η οποία ήταν ε, η πιο οραματική δήλωση στην ιστορία. Οι αλλαγέ ήταν εξαιρετικά βραδίες. Ε, ε, στο ΙΕ έχουμε την ευκαιρία να αξιολογήσουμε ε, αυτή την συνδιάσκεψη. Η πορεία ήταν βραδία γιατί υπάρχει μυθιστολογικό και συνταξιοδοτικό χάσμα. μικρά ποσοστά, χαμηλά ποσοστά απασχόληση για τις γυναίκες, λίγες για τις γυναίκες σε υψηλές θέσεις ε, άσκηση βίας κατά των γυναικών κλπ. Γι' αυτό θα πρέπει να προβούμε στο πλαίσιο της Συνόδου σε μια κοινή δήλωση. Το 2021 θα είναι κρίσιμο έτος. Όλοι φέρουμε ένα μερίδιο της ευθύνη. Δεν μπορούμε να απιστοδρομήσουμε. Όλοι έχουμε συλλογική για ατομική ευθύνη. Θα ήθελα να σας πω ότι η περιβαλλοντική βιωσιμότητα είναι θεμελιώδης για τον πλανήτη, αλλά επίσης και, για την, και η βιωσιμότητα ε, και η ισότητα των δύο φύλων. Ευχαριστώ πολύ. Οι γυναίκες είναι ε, στην, ε, στο περιθώριο της κοινωνίας ε, σε πολλές χώρες. Έχουν επίσης κακή πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης και γενικότερα η ζωή τους είναι πιο υποβαθμισμένη. Αυτό πολλές φορές αποσιωπάται. Ε, καμιά φορά στα νοσοκομεία, ε, ειδικέ ομάδες, ε, ιδιαίτερες ομάδες γυναικών απομονώνονται και δεν τους προσέχει το ιατρικό προσωπικό. Επίσης, πολλές φορές θυρώνονται χωρίς την, ε, στην κατάθεσή τους. Η, καλή, η Σλοβακία ε, να προβλέψει αποζημίωση για τις θυρωμένες γυναίκες. Ε, ε, μέχρι τώρα, μετά από 14 χρόνια, μία μόνο γυναίκα αποζημιώθηκε. Θα πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τις γυναίκες από ε, ειδικέ ομάδες. Πώς θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματά τους. Η κυρία Καρβάλιο, ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, να πούμε κάτι θεμελιώδες που, που υπάρχει και στο χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων και στην, στο χάρτη του ΟΗΕ και πρέπει να είναι ε, βασική και για την πολιτική της Ένωσης και την εξωτερική πολιτική. Είναι ε, θα πρέπει στη Νέα Υόρκη να ε, επιτύχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα διότι πρέπει να είμαστε αρμόδιοι ε, και επί της ουσίας όταν προασπίζουμε τα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών και την ισότητα των φίλων. Θα πρέπει να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη των δικαιωμάτων αυτών. Ήδη είμαστε ε, προχωρημένοι σε θέματα χειραφέτηση, δημιουργίας ίσων ευκαιριών για τις γυναίκες και τα κορίτσια σε όλους τους τομείς. Ελπίζω ότι θα έχουμε δεσμεύσεις ε, ε, θετικές για να εφαρμόσουμε όλα τα μέτρα μας και το 2003 να εφαρμόσουμε τους στόχους της χιλιετίας. Ακολουθεί το Catch the Eye. Ο κύριος Κύριε Επίτροπε, ελπίζω ότι αυτή η νέα στρατηγική θα γίνει πραγματική επανάσταση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και όχι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει να συνοδευτεί από συγκεκριμένα και δεσμευτικά και υποχρεωτικά μέτρα. Νομίζω ότι θα πρέπει επίσης να φτιάξουμε και μια ευρωπαϊκή οδηγία για το θέμα αυτό. Λυπάμαι όμως για το γεγονός ότι είναι ελάχιστοι ευρωβουλευτές στην αίθουσα. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον δηλαδή για αυτό το θέμα μια υγιής λύση θα ήταν να υιοθετήσουμε ευρωπαϊκά μέτρα, ευρωπαϊκή λύση. Και ελπίζω τα δικαιώματα και υποχρεώσεις να είναι η ίδια για όλους και όλες. Σας ε, ενθαρρύνω να συνεχίσετε προς την ίδια ατραπό. Η κυρία Σαρντόνε, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Πριν από λίγους μήνες, στο Ιράν, καταδικάστηκε μια γυναίκα δικηγόρος που υπερασπιζόταν τα δικαιώματα των γυναικών. Γυναικών που δεν ήθελαν να βάλουν ε, το... Ε, να βάλουν ε, να καλύψουν το, πρόσωπό τους. Και καταδικάστηκε σε 148 βουρτουλιές και πολλά χρόνια φυλάκισης. αλλά και μία 15χρονη εδώ στην Ευρώπη ε, εδάρι από τους γονείς της γιατί ήθελε να, βάλει, να καλύψει το κεφάλι της. Ε, ένα κοριτσάκι επίση, ε, επειδή έκανε, ζέστη δεν ήθελε να βάλει τίποτα στο κεφάλι του και οι γονείς του το έδιραν. Επίσης άλλα κορίτσια τα οποία περιφέρονταν με σορτσάκια τιμωρήθηκαν. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μιλάει για τις προτεραιότητες σε αυτή την 24η Σύνοδο του ΟΗΕ για την κατάσταση και τη θέση των γυναικών. Εμένα θα μου άρεσε η Ευρώπη να σταματήσει αυτή την υποκρισία. Που, υποκρισία που την κάνει να αποστρέφει το βλέμμα. Δεν βλέπει ότι κάποιες συμπεριφορές συνδέονται με μια συγκεκριμένη κουλτούρα και με μια συγκεκριμένη θρησκεία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Τόμασιτς για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. το ε, μοντέλο ισότητα των φίλων που έχουμε στο δυτικό κόσμο δεν υπάρχει και στου υπόλοιπου πολιτισμού και κουλτούρε ανά τον κόσμο. Θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε τα παγκόσμια φόρα και ό,τι δυνατότητα μα προσδίδει ο ΙΕ για να προωθήσουμε τα δικαιώματα των φίλων και την ισότητα. Ε, σε κάποιε κουλτούρε οι γυναίκε βρίσκονται σε τόσο. Ε, θέση που οι κοινωνίες Πραγματικά πολλές φορές τις ε, εξαναγκάζουν σε άμβλωση αν περιμένουν κορίτσι. Τα κορίτσια δεν έχουν καν δικαίωμα να γεννηθούν σε αυτές τις κουλτούρες. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε ε, κάθε δυνατή προσπάθεια για να αντιμετωπίσουμε τέτοια φαινόμενα. Στην ε, σύνοδο του ΙΕ θα πρέπει να καταπολεμήσουμε αυτήν την απαράδεκτη πρακτική της ε, δολοφονίας αγέννητων κοριτσιών που είναι τόσο διαδεδομένη σε κάποιες χώρες. Και τώρα καλώ την ε, Υπουργό Μπρνιέτ να μιλήσει εκ μέρους του Συμβουλίου, της Προεδρίας του Συμβουλίου. Ευχαριστώ, αξιότιμοι κύριοι Βουλευτέ. Πρόκειται για την 24 ε, η Σύνοδο για την ε, γυναίκα. Έχουμε βάλει ψηλά τον πύχη και από νωρί υποσχεθήκαμε προς όλες τις χώρες ότι θα έχουμε ανοιχτό πνεύμα. Θέλουμε να υπάρξει συνένεση, να προβούμε σε κάποια διακήρυξη και δήλωση συγκεκριμένη. Οπότε να προχωρήσουμε μετά σε ανάληψη δράση σε σχέση με αυτή την συνάντηση. Θέλουμε να ε, επαληθεύσουμε το ότι είμαστε προσιλωμένοι στην πλήρη ισότητα και ότι θα πρέπει γυναίκες και ανήλικες γυναίκες να απολάβουν όλων των δικαιωμάτων τους. Και είναι κρίσιμος ο ρόλος των θεσμικών οργάνων. Είμαστε περήφανοι που προς τα εκεί κινείται το Συμβούλιο προς μια ισότητα των δύο φύλων στην Ευρώπη. Και προσδοκούμε σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο στο μέτωπο αυτό. Σας ευχαριστούμε που είσαστε τόσο δυναμικοί και έχετε ψηλά στο θεματολογιό σας το εν λόγω ζήτημα. Σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε κυρία Υπουργέ. Κλείνει εδώ η συζήτηση για το ζήτημα τούτο. Έχουμε δύο προτάσεις για ψηφίσματα σε σχέση με αυτήν ε, την συζήτηση. Ένα κοινό ψήφισμα από Σοσιαλδημοκράτες Πράσινους, Renew, Γκουε και ΕΛΚΑ. Και χωρίς την πρόταση από το ECR η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο. I uh, Έχω μία ανακοίνωση πριν αρχίσουμε την επόμενη συζήτηση. Το ΕΛΚ και το ID έχουν κοινοποιήσει απόφαση να αλλάξουν κάποιοι διορισμοί βουλευτών σε αντιπροσωπείες κλπ και αυτά θα καταχωριστούν στα πρακτικά της σημερινής ε, συνεδριάσεως ε, με χρόνο την ώρα ε, αυτής της ανακοινώσεως. Το επόμενο θέμα σήμερα σε διάταξη είναι η έκθεση τσόλα που αφορά τα γνήσια και πλαστά έγγραφα σε σχέση με το μητρό στο ίντερνετ. Σας υπενθυμίζω τις οδηγίες για χρήση ηλεκτρονικής κάρτας. Αυτές βρίσκονται στην είσοδο του ημικυκλίου. Σας υπενθυμίζω ότι μπορείτε να υποβάλλετε ε, ερωτήσεις με μπλε κάρτα μόνο αφού ολοκληρωθούν οι αγορεύσεις των εκπροσώπων των πολιτικών ομάδων. Η κυρία Μετσόλα είναι η πρώτη συνάδελφος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ήταν ε, μακρύς ο δρόμος για να φτάσουμε στο αποτέλεσμα στο οποίο έχουμε καταλήξει πλέον. Η παραποίηση ε, εγγράφων υποσκάπτει την ασφάλεια ε, του χώρου Σέγγεν, ένας χώρο όπου υπάρχει ελεύθερη κυκλοφορία χωρίς συνοριακούς ελέγχους. Αυτή η νέα νομοθετική πράξη αντιμετωπίζει το πρόβλημα, εξασφαλίζοντας ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρών εταίρων όσον αφορά την, τον εντοπισμό γνήσεων και πλαστών εγγράφων. Με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλιστεί η ασφάλεια των εξωτερικών μας συνόρων και κατ' επέκταση των πολιτών που εκπροσωπούμε, ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε να απολαμβάνουμε τα δικαιώματα και τα ωφέλη του χώρου Σέγγεν. Αλλά για να γίνει αυτό βεβαίως πρέπει να υπάρχει μια αποτελεσματική διαχείριση των εξωτικών ε, συνόρων. η νομική αυτή πράξη αποτελεί συστατικό στοιχείο μια τέτοια στρατηγική, καθώ η διασφύλαξη των συνόρων και η καταπολέμηση τη εγκληματικότητα θα μα βοηθήσει να προσδιορίσουμε και να εντοπίζουμε τα πλαστά έγγραφα. θεσπίζεται ένα νέο πλαίσιο το οποίο προβλέπει την ε, συνεργασία και της Frontex καθώς και όλων των ε, συμμετεχόντων κρατών μελών που θα ενημερώνονται και θα εκπαιδεύονται για το πώς μπορούν να εντοπίζουν και να ταυτοποιούν πλαστά έγγραφα. Προσδιορίζεται ο ρόλος ε, της, του Frontex όσον αφορά τη διαμόρφωση αυτού του συστήματος FADO και το φάντο αυτό πλέον θα συμπεριλαμβάνει περισσότερες πληροφορίες από αυτές που σήμερα ε, συλλέγονται σε σχέση με τα γνήσια και τα πλαστά έγγραφα. Με κεντρική διαχείριση. Ο Frontex θα πρέπει επίσης να έχει την ευελιξία να αναβαθμίζει ε, το σύστημα Φάντο. Σύντομα επίσης θα, ε, δημοσιευθούν και κατευθυντήρες γραμμές για το πώς καλύτερα μπορεί κανεί να εντοπίζει πλαστά έγγραφα. Έχουμε κάνει ό,τι περνούσε από τα χέρια μα, ώστε βεβαίω πάντοτε να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα. Το αποτέλεσμα που επιδιώκουμε είναι περισσότερη ασφάλεια και προστασία και ταυτόχρονα εγγύηση ε, της ε, ασφάλειας των πολιτών, που είναι απαραίτητο στοιχείο στην, ε, στον ε, αγώνα, στην καταπολέμηση των πλαστών εγγράφων στο Σέγγεν είναι κρίσιμο να υπάρχει μια τέτοια δυνατότητα ελέγχου των πλαστών εγγράφων ως ε, τρόπος για τη διαφύλιξη των εξωτερικών ε, συνόρων. Μπορεί το σύστημα αυτό να φαίνεται εκ πρώτης όψεως ε, ως ιδιαίτερα τεχνικό, όμως θεωρώ ότι είναι απαραίτητο στοιχείο για τη διαφύλαξη των εξωτερικών μας συνόρων. Η ευθύνη υπό τον κανονισμό αυτό έχει διευρυνθεί μετά από δικές μας προσπάθειες. Καταγράφονται και παρατίθενται ακριβώς οι αρμοδιότητες όλων των οργανισμών και των κρατών μελών και ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων θα εξασφαλίζεται πάντοτε με βάση το ευρωπαϊκό δίκαιο. Επίσης εξασφαλίσαμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχει περισσότερο λόγο όσον αφορά το φάντο. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω το Συμβούλιο, την Φιλανδική και την Κροατική Προεδρία, καθώς και τους συναδέλφους μας, συναδέλφους μου για την επικοδομητική και συναδελφική τους ε, στάση. Προσβλέπω στην ε, συζήτηση που θα κάνουμε σήμερα εδώ στην Ολομέλεια και περιμένω να μου δώσετε το λόγο για τις καταληκτικές μου παρατηρήσεις. Ευχαριστούμε κυρία Συγγήτρια. Η κυρία Ντάλη έχει το λόγο εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ κυρίες και κύριοι βουλευτές, ευχαριστώ για αυτή τη συζήτηση. Οι πολίτες μας θεωρούν την ασφάλεια ως μία από τις πρώτες προτεραιότητες και τα πράγματα που τους ανησυχούν. Περιμένουν να κάνει κάτι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ασφάλεια και η ελευθερία πάνε χέρι-χέρι. Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα χώρο ασφαλείας για όλους τους Ευρωπαίους. Το να είναι κανείς ασφαλής είναι αναγκαίο και αναγκαία προϋπόθεση για να μπορεί να ζει, να απολαμβάνει των δικαιωμάτων του, να ε, ζει, να σπουδάζει και είναι και απαραίτητο για την οικονομία. Ο καθένας που βρίσκεται στην Ευρώπη έχει το δικαίωμα ως άνθρωπος να είναι ασφαλής. Ε, το βαρόμετρο, το ευρωβαρόμετρο για την κυβερνοασφάλεια του 2019 δημοσίευσε πρόσφατα απορίσματα που δείχνουν ότι το 2, τα δύο τρίτα των ε, όσων απήντησαν στο ερωτηματολόγιο ανησυχούν μήπως πέσουν θύματα ε, κατάχρησης της ταυτότητάς τους ή κλοπής της και μια εύρυθμη περιοχή, ένα εύρυθμο χώρο του Σέγγεν με την ε, ελεύθερη κυκλοφορία απαιτεί καλό έλεγχο στα εξωτερικά σύνορα. Πρέπει να κάνουμε αποτελεσματικό έλεγχο και να ε, βλέπουμε ποιοι ε, περνάνε τα εξωτερικά σύνορα προ όφελο όλων μα. Η ανάγκη για ενίσχυση τη εσωτερική μας ασφάλεια στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει οδηγήσει στην έγκριση μια σειρά από πρόσφατες νομοθετικές πράξεις, όπως για παράδειγμα τα, το σύστημα για, την Ευρωπα... για τα ευρωπαϊκά ταξιδιωτικά έγγραφα και την εξουσιοδότηση, το σύστημα διαλειτουργικότητας μεταξύ των ευρωπαϊκών ε, συστημάτων πληροφοριών και το νέο κανονισμό για την Ευρωπαϊκή Φυλακή και Ακτοφυλακή. Σήμερα έχουμε ένα επιπλέον παράδειγμα που είναι τα γνήσια και πλαστά έγγραφα και το σύστημά τους ε, στο διαδίκτυο. Μια νέα βάση δεδομένων που θα υποστηρίζει τα κάτι μέλη ώστε να εντοπίσουν γνήσια ή πλαστά έγγραφα. Ευχαριστώ ε, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ε, για την επικοδομητική τους εργασία σε αυτή την τελική συμβαστική λύση πραγματικά ε, προσφέρουμε θέμενη αξία. Οι διάφορες, ε, το, νέο σύστημα, το ΦΑΝΤΟ, είναι πολύ χρήσιμο για την ακτοφυλακή και τη συνοροφυλακή όταν κάνουν ελέγχου στα σύνορα. Και πραγματικά παράσχει πληροφορίε στι αρχέ των κρατών μελών για τι νέε μεθόδου και για τα νέα γνήσια έγγραφα που μπορεί να κυκλοφορούν χρησιμοποιούνται χιλιάδες περιγραφές γνησίων εγγράφων, εκατοντάδες πλαστών οι οποίες καλύπτουν περισσότερα έχουν να κάνουν με 30 ε, χώρες που συμμετέχουν και 130 οργανισμούς ε, διεθνώς. Ε, εντοπίζονται απόπειρε κλοπής ταυτότητας για υπεξαίρεσης ταυτότητας για σκοπούς λαθρομετανάστευσης. Η τελική πολιτική συμφωνία θα βελτιώσει έτσι περαιτέρω την λειτουργία του συστήματος γνήσεων και πλαστών εγγράφων στο διαδίκτυο και θα επιτρέψει να μεταφερθεί η ε, διαχείρισή του στην Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή. Η ασφάλεια είναι κορυφαία ανησυχία και μέρημνα των Ευρωπαίων πολιτών. Περιμένουν αποτελέσματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να αισθάνεται και να είναι πράγματι ε, προστατευμένος οι απειλέ που προέρχονται από το οργανωμένο έγκλημα, την τρομοκρατία και την αγορά των ναρκωτικών δηλητηριάζουν τι κοινωνίε μας. Γι' αυτό ακριβώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναγγείλει μια νέα στρατηγική ασφαλείας της Ευρωπαϊκή Ένωση, για το δεύτερο τρίμηνο φέτο, και ως μέρος της στρατηγικής αυτής για την εσωτερική ασφάλεια θα δώσουμε προτεραιότητα σε τρει ε, τομεί προτεραιότητα. Το οργανωμένο έγκλημα που συμπεριλαμβάνει τα ναρκωτικά, τα, πυρομαχα, τα, πυρομαχ, ε, τα πυροβόλα όπλα την ε, αγο... πορεία ναρκωτικών και ανθρώπων, την τρομοκρατία και τη ριζοσπαστικοποίηση και την καταπολέμηση των ε, εγκληματικών ενεργειών στην ψηφιακή εποχή. Για να υποστηρίξουμε το χώρο ελεύθερη κυκλοφορία που είναι ένα από τα σύμβολα τη Ένωσή μα, θα πρέπει να προωθήσουμε αυτά τα νέα στοιχεία και το νέο σύμφωνο τη μετανάστευση, όπω έχει ανακοινωθεί στι νέε πολιτικέ κατευθυντήριε γραμμέ τη Προέδρου Φόντερ Λάιεν. Ε, υπ' αυτήν την έννοια η επίκαιρη υλοποίηση όλων των νέων συστημάτων πληροφοριών θα είναι ε, απότατος στόχος της σφαιρικής προσέγγισης της μετανάστευσης. Θα επικεντρωθούμε στα εξωτερικά σύνορα το ίδιο όσο και στην εσωτερική ασφάλεια, καθώς και την ισχυρή και ανθεκτική επεξεργασία των στοιχείων. Θα πρέπει να προωθήσουμε τους νομικούς διάβλους και την, ε, να καλλιεργήσουμε την καλύτερη ένταξη στις κοινωνίες μας. Σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας και προσβλέπω στην συζήτηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Τώρα έχουμε τους αγορητές ε, από τις πολιτικές ομάδες και ξεκινούμε με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Κύριε Ράντεφ, έχετε ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, η απάντηση σχετικά με τα έγγραφα είναι κάτι το οποίο υπονομεύει την ασφάλεια στην περιοχή Σέγγεν, εκεί που δεν υπάρχουν συνορικοί έλεγχοι. Τα παραπημένα πλαστά έγγραφα χρησιμοποιούνται συχνά από αλλοδαπού οι οποίοι αναζητούν μια καλύτερη ζωή στην Ευρώπη. Και αυτά τα έγγραφα μπορεί να αποκτώνται έναντι 5 ή 6 ευρώ. Και όμως τα χρησιμοποιούν οι, ε, το οργανωμένο έγκλημα και οι τρομοκράτε. Επίση, και όσοι ε, κάνουν εμπόριο όπλων και αυτοί οι οποίοι εμπορεύονται ε, κλεμμένα αυτοκίνητα. Τα γνήσια έγγραφα πάρα πολλές φορές εκδίδονται επί τη βάση ψευδών ε, στοιχείων, ταυτότητος. Αυτό κάνει πιο δύσκολη την κατάσταση του εντοπισμού και είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουν ασφάλεια τα αξιωτικά έγγραφα και επίσης να γίνεται έτσι κάποιο είδους διαχείριση της υποδομής για αυτά τα έγγραφα. Από την άλλη μεριά η συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων αρχών θα πρέπει να γίνει ε, πιο εντατικά σε συνεργασία και με τις διοκτικές αρχές και θα πρέπει να υπάρχει επαφή μεταξύ των ε, ε, εκδιδουσών αρχών και των διεθνών θεσμικών οργάνων. Σε αυτό το πλαίσιο παρακαλώ να εγκρίνετε αυτή την πρόταση και το σύστημα φάντο να εγγραφεί, να ενταχθεί μάλλον στο σύστημα που έχουμε ε, και έτσι να ολοκληρωθεί η σχετική μεταρρύθμιση του συστήματος. Ο κύριος Λόπεθ Αγγιλάρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε Ντάλη. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν την ευθύνη, έχουν και το δικαίωμα να ελέγχουν ποιο μπαίνει στην περιοχή ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων του Σέγγεν. Όμω, αναδύεται ένα πρόβλημα το ότι έχουμε πολλαπλασιασμό, αύξηση των ε, παρατημένων και πλαστών εγγράφων σε σχέση με την ταυτότητα του προσώπου. Αυτό είναι κακό για την ασφάλεια, διότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε έγκλημα, σε ξέπλυμα χρήματο και διάφορες άλλες παράνομες πράξεις, αλλά ακόμα και σε τρομοκρατικές πράξεις. Θα πρέπει κάτι να κάνει το Κοινοβούλιο και το έχει πει και σε σχέση με τη διαδικασία ασύλου χρειάζεται κάτι το οποίο έχει σχέση με την αποθήκευση, την ανταλλαγή δεδομένων ε, σε σχέση με τα έγγραφα για να καταπονηθούν οι σχετικές απάτες. Οπότε θα πρέπει ο κόσμος να δείχνει εμπιστοσύνη προς ε, τις υπηρεσίες ε, φύλαξης συνόρων, ε, και την ακτοφυλακή. Ε, εγκρίναμε ένα σχετικό νομοθέτημα το 19, ούτως ώστε να υπάρχει ανταλλαγή των σχετικών πληροφοριών με τρόπο ασφαλή. Να εμπλέγονται δηλαδή όλες οι αρχές οι οποίες είναι συναρμόδιες και έτσι να λαμβάνεται υπόψη η αληθή ταυτότητα των προσώπων που δικαιούνται την ελεύθερη κυκλοφορία στο χώρο Σέγγεν. Εμείς ανέκαθεν θέλουμε αυτό να είναι συμβατό με τα όσα έχουμε κάνει για να υπάρχουν εγγύησει όσον αφορά την εμπιστευτικότητα των δεδομένων, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και βέβαια τι ε, αρχέ που είναι θεμέλιε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για το δικαίωμα του να ε, καταπολεμάται ε, η, η ανασφάλεια και όλοι να μπορούν να κυκλοφορήσουν και να έχουν στη διάθεσή του αυτά τα τεχνολογικά εργαλεία που χρειάζονται. Αλλά να υπάρχει και ασφάλεια δικαίου που χρειάζεται. Επίση, να υπάρχει και διαλειτουργικότητα σε σε σχέση με αυτά τα συστήματα των δεδομένων ε, και βέβαια να είναι όλα αυτά συμβατά με τον χάρτη των δικαιωμάτων. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εκ μέρους του Ρινιού, ο κύριος chair. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχά, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Ρομπέρτα Μετζόλα, την εισηγήτρια, για το έργο τη. Ω νέο Ευρωβουλευτή, που εργάζομαι ε, επί του πρώτου νομοθετικού φακέλου, νομίζω ότι η ηγετική της ικανότητα ήταν προφανής. Τώρα, επί της ουσίας, ε, το σύστημα που ε, έχουμε στην διάθεσή μας για την, τον εντοπισμό γνήσεων και πλαστών εγγράφων εδώ και πολλά χρόνια δέχεται τεράστιες πιέσεις λόγω του όγκου των εισερχόμενων και εξερχόμενων ανθρώπων. Για την ε, ε, ε, ο εντοπισμός πλαστογραφημένων εγγράφων αποτελεί μεγάλη πρόκληση για τις αρχές μας. Το σύστημα Φάντο βρίσκεται σε ισχύ εδώ και κάποια χρόνια. Πλέον θέλουμε από διακυβερνητικό σύστημα να γίνει κοινοτικό σύστημα ώστε να μπορέσει να ενταχθεί στο ευρύτερο νομοθετικό πλαίσιο ε, του ευρωπαϊκού δικαίου. Αυτό θα ενισχύσει την εξασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και θα ε, ε, ενισχύσει τις εγγύσεις όσον αφορά την πρόσβαση στα δεδομένα αυτά. Με αυτόν τον τρόπο η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων θα γίνεται μόνο εκεί όπου πραγματικά είναι απαραίτητη για τον σκοπό της διερεύνησης ή του εντοπισμού πλαστών εγγράφων. Επίσης πλέον υπάρχουν κανόνες για τα κράτη-μέλη, τα οποία θα πρέπει να καθορίζουν ποιες ακριβώς αρχές θα έχουν πρόσβαση στο σύστημα ΦΑΝΤΟ, ποιο θα είναι το επίπεδο της πρόσβασης και πότε θα πρέπει να κοινοποιούνται οι σχετικές ενέργειες προς την Κομισιόν. Η ΔΕ Κομισιόν θα πρέπει να ενημερώνει πάντα το Κοινοβούλιο. Έτσι, συνολικά θα εξασφαλίζεται καλύτερα η διαφύλαξη των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης και η επιβολή του νόμου. Γι' αυτό και καλώ τους ε, ευρωβουλευτές συναδέλφου μου να υποστηρίξουμε το κείμενο αυτό. Ευχαριστούμε. Εκ μέρου ε, του ID, ο κύριος Ταρντίνο. Η κυρία Ταρντίνο. Ευχαριστώ ε, πρόεδρε. Ευχαριστώ τη συνάδελφο για τη δουλειά της. Εδώ έχουμε πολλές απάτες που έχουν ε, καταγραφεί στο χώρο Σέγγεν τα τελευταία χρόνια. Επειδή τα γνήσια έγγραφα δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τα πλαστά. Ο παρόν κανονισμός μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε ένα σύστημα για τη διάκριση στο διαδίκτυο των ε, πλαστών από τα γνήσια έγγραφα και να χρησιμοποιείται αυτό και από το Frontex. Η εσωτερική ασφάλεια και προστασία που μας ζητούν οι πολίτες μας μας επιβάλλει να έχουμε ένα διαρκές επίπεδο εντοπισμού των ε, πλαστών εγγράφων και αυτό να είναι διαρκές διότι χρησιμοποιούνται για, πολλές, ε, για πολλούς σκοπούς ε, έγγραφα όπως για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ή για τρομοκρατικούς σκοπούς ή για την ελαφρομετανάστευση. Πολύ συχνά χρησιμοποιούνται από ετούντες άσυλο που προσπαθούν να μπουν στην Ευρώπη τα έγγραφα αυτά. Πρόκειται για συμπεριφορές τις οποίες δεν μπορούμε να δεχτούμε και πρέπει να πάυσουν. Θα πρέπει η αστυνομία αστυνομία, η συνοροφυλακή και οι τρονικέ αρχέ να έχουν μια τέτοια βάση δεδομένων που να του επιτρέπει να εντοπίσουν γρήγορα τα πλαστά έγγραφα και να αναχαιτήσουν τα σχετικά φαινόμενα. Για αυτού του λόγου στηρίζουμε την πρόταση, παρόλο που διαφωνούμε με το ότι κάποιοι ιδιώτε θα έχουν και εκείνη πρόσβαση στο φάντο, έστω και σε συγκεκριμένε και υπό συγκεκριμένε προποθέσει. Πάντω, με την αναθεώρηση του, οργανισμού, της, του οργανισμού Frontex, θα πρέπει να κοιτάξουμε το φάντο να χρησιμοποιείται αποτελεσματικά στην αναχέτηση της απάτης από τις αρχές των κρατών μελών. the Ευχαριστούμε από τους Πρασίνους η κυρία Μπρικμό. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ συνάδελφοι για την καλή συνεργασία στο θέμα αυτό. Είναι ένα ντοσχέ πολύ τεχνικό που ζητά ε, την αλλαγή στη διασύνδεση των βάσεων δεδομένων. Δυστυχώ αυτή την διαχείριση την αναλάβει πλέον η Frontex. Θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ για να μην ενισχυθεί η εντολή του οργανισμού πλαγίου, διότι το ΦΑΝΤΟ δεν είναι ένα εργαλείο καταπολέμηση τη λαθρομετανάστευση. Είναι, κατα... κατά της είναι για την καταπολέμηση τη πειρατεία τη παραπίση εγγράφων. Θα πρέπει λοιπόν να προβλέψουμε εγγύσει ώστε τα τρίτα μέρη, αεροπορικέ εταιρείε, ιδιωτικέ εταιρείε να μην έχουν ε, απεριόριστη πρόσβαση, αλλά περιορισμένη στη βάση των δεδομένων. Θα περιέχει και προσωπικά δεδομένα η βάση δεδομένων, οπότε θα πρέπει να μην μπορεί να υπάρξει ταυτοποίηση μέσω των εγγράφων του Φάντο. Ε, επίσης, θα παρακολουθούμε προσεκτικά την δημοσίευση των διαφόρων ε, κατεξουσιοδότηση πράξεων. Ευχαριστώ. Για τους μεταρρυθμιστές συντηρητικούς έχει το λόγο ο κύριος Μπούσαντε Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχουμε χιλιάδες τέτοια έγγραφα στα εξωτερικά μας σύνορα κάθε χρόνο. Το 18, σύμφωνα με την Frontex, είχαμε 7.000 αλλοδαπούς οι οποίοι εμφανίστηκαν με πλαστά έγγραφα και θέλανε να περάσουν τα σύνορα της Ένωσης. Έχουμε πολλές μεθόδους ε, πλαστογράφησης. Ε, πρόκειται πραγματικά για κάτι πολυχρηστικό, για ξέπλυμα χρήματος, για τρομοκρατία και τέλος πάντων για παράνομη εισόδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε αναδεικνύεται το πόσο σημαντικό είναι να προστατεύσουμε τα σύνορα και να έχουμε έλεγχο της μετανάστευσης. Όλα αυτά σημαντικά για την ασφάλεια των Ευρωπαίων. Οπότε το σύστημα Φάντο ε, θα αξιοποιήσει την ε, εμπειρία της Frontex. Θα έχουμε ταχεία ανταλλαγή στοιχείων. Βέβαια τα κράτη-μέλη ε, μπορούν να κάνουν καλύτερα, μπορούν να κάνουν περισσότερα πράγματα για την δίωξη των εγκλημάτων. Η πολιτική μας ομάδα προβληματίζεται ε, με αυτά τα οποία γίνονται ε, όσον αφορά τον, την είσοδο των αλλοδαπών. Εμείς θα ψηφίσουμε υπέρ. Ο Πρόεδρος. Για την ΚΟΕ έχει τον λόγο η κυρία Σύρα Ρέγκο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα πρέπει να θυμηθούμε ότι την εποχή του φασισμού στην Ευρώπη ήταν χιλιάδες αυτοί, ήταν υποχρεωμένοι να χρησιμοποιήσουν πλαστογραφημένα έγγραφα για να γλιτώσουν και αυτό. Ε, έχει συζητηθεί ε, και δεν είναι μόνο θέμα τεχνοκρατικό όπως συζητούμε τώρα για αυτά τα μέτρα. Πρόκειται για το ζήτημα των αυθεντικών και των πλαστών εγγράφων. Δεν θέλουμε την Ευρώπη φρούριο. Έχουμε χιλιάδες ε, μεταναστών που χρησιμοποιούν τέσσερα εγγράφα. Αυτό έρχεται κόντρα στα όσα ε, προβλέπει η Σύμβαση της ε, Γενέβης για το ποιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν ταξιδιωτικά έγγραφα. Θέλουμε να θωρακίσουμε την Ευρώπη, να την κάνουμε φρούριο, να την κάνουμε γέφυρα εκδίωξης και, και, και έκδοση προσώπων θα πρέπει να έχουμε κάποιο είδους θεωρήσεις ανθρωπιστικές σε σχέση με την προέλευση κάποιου και θα πρέπει οπωσδήποτε να αναγνωριστούν οι κλιματικοί πρόσφυγες. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε. Τώρα ολοκληρώνονται οι αγορτές των πολιτικών ομάδων και στο εξή θα έχουμε ε, ερωτήσεις με μπλε κάρτα. Θα επιτρέπονται. Ο επόμενος αγορητής είναι ο κύριος Λέναρς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι πολύ καλό το σύστημα για να μπορέσουμε να εντυπίσουμε τα πλαστά έγγραφα. Η Frontex ε, μπορεί να προστατεύσει καλύτερα το χώρο Schengen και καλό θα ήταν να βαθμιστούν οι δυνατότητές της. Βεβαίω η ασφάλειά μα θα βρίσκεται πλέον επιγραμμικά ε, στο διαδίκτυο. Γι' αυτό και οι αρχέ θα πρέπει να μπορούν να διαπιστώσουν κατά πόσον τα έγγραφα είναι γνήσια ή όχι. Χρειάζονται συγκεκριμένε ε, συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και ε, ρυθμίσεις που να είναι ξεκάθαρα για όλους. Να γνωρίζουν όλοι σε κάθε χώρα τι είναι νόμιμο και τι όχι. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να μπορούν να είναι βέβαια ότι είναι πάντοτε επικαιροποιημένες και διαθέσιμες 24 ώρες 24 ώρες 7 μέρες την εβδομάδα. Το νέο σύστημα ε, είναι ευπρόσδεκτο και θα είναι κέρια σημασίας, διότι η ασφάλεια και η γνησιότητα των εγγράφων πάνε χέρι-χέρι. Ευχαριστώ λοιπόν τον συγητή και προσβλέπω σε ένα σύστημα που θα λειτουργεί καλύτερα για τον ε, νέο ψηφιακό κόσμο. Ευχαριστούμε. Η κυρία Κινίτσι, για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η καταπολέμηση των πλαστών εγγράφων και η κυκλοφορία του στον χώρο Σέγγεν ε, είναι προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ των αρχών και ε, στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Για να υπάρχει δραστική ε, καταπολέμηση όμως θα πρέπει να υπάρχει και σωστή ανταλλαγή των πληροφοριών, κάτι που δεν μπορεί να γίνεται μόνο μεταξύ των αρχών των κατων μελών, αλλά πλέον με τις απαραίτητες εγγυήσεις θα γίνεται και μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των αρχών των τρίτων χωρών ιδιωτικέ εταιρείε όπω οι αεροπορικέ, που θα μπορούν να επιτρέψουν την να ενισχυθεί η εύρυθμη λειτουργία του συστήματο Φάντο. Τα στοιχεία τη Europol μα δείξαν ότι πολλέ φορέ τα πλαστά έγγραφα ε, εξυπηρετούν τη λειτουργία των ε, ομάδων οργανωμένων εγκλήματο για σοβαρά εγκλήματα όπω την λαθρομετανάστευση, την εμπορία ανθρώπων ή την προετοιμασία τρομοκρατικών δράσεων, την εμπορία, το διακίνηση ναρκωτικών. Γι' αυτό λοιπόν μεταξύ άλλων χρειάζεται καλύτερος έλεγχος στα εξωτερικά σύνορα. Είμαστε υπέρ του να μεταφέρει ο κανονισμός την αρμοδιότητα για τη διαχείριση των ε, ε, ε, πλαστών και γνησίων εγγράφων από το Συμβούλιο στη Frontex και να μπορεί να βελτιωθεί η εντολή του οργανισμού αλλά με τη σωστή εφαρμογή ώστε να είναι αποτελεσματικοί οι κανόνε που έχουν εγκριθεί ω τώρα. Ευχαριστώ τη συνάδελφό Μετσόλα για τη δουλειά που έχει κάνει και εύχομαι ο κανονισμός αυτός πραγματικά να εγκριθεί ε, με ευρία πλειοψηφία από το Κοινοβούλιο. Ευχαριστούμε κύριε Προκατσίνη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η συμφωνία ε, θα είναι εφόσον εγκριθεί αρκετά τεχνικού χαρακτήρα, έχει όμως και πολιτικό νόημα κατά δύο τρόπους. Πρώτον, η απάτη μέσω των εγγράφων είναι μια μεγάλη απειλή για όλους μας Και η συνεργασία μεταξύ 100 μελών, αυτή που ζητά το σύστημα Φάντο, θα είναι πραγματικά ε, επιτυχία εφόσον την ε, ολοκληρώσουμε θα πρέπει να ε, λειτουργήσει βεβαίω εύρυθμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να μην γίνει εργαλείο που θα εξυπηρετεί του σκοπού κάποιων. Κάτι άλλο που θα πρέπει να σκεφτούμε είναι ε, η ελαχιστοποίηση των δεδομένων που θα πρέπει να δούμε τον ορισμό τη. Οι περιορισμοί που προβλέπονται για την ανάκτηση προσωπικών δεδομένων είναι μια χαμένη ευκαιρία για να καταπολεμήσουμε αποτελεσματικά το οργανωμένο έγκλημα και την λάθρο μετανάστευση, την παράτυπη μετανάστευση. Ε, η αριστερά αυτού του κοινοβουλίου άλλωστε έχει δείξει ότι είναι απομακρυσμένη από την πραγματικότητα με τις προτάσεις της εδώ. Ο κύριος Δεχόφσκι, ναι. Eh, ναι, ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Κυρία Επίτροπε, κυρία Εισηγήτρια, σας ευχαριστώ για την εξαιρετική δουλειά που έχετε κάνει. Το 2015 εγώ βρέθηκα στα σύνορα μεταξύ Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας. Τότε είχαν συγκεντρωθεί 55 διαφορετικά συριακά διαβατήρια, εκ των οποίων κανένα δεν ήταν γνήσιο. Πολλοί άνθρωποι κατέληξαν στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πλαστά έγγραφα. Γι' αυτό και είναι τόσο σημαντικό και η συγκεκριμένη πρόταση κανονισμού, διότι ενώ εμφανίζεται ως ένα τεχνικό εργαλείο, στην πραγματικότητα έχει μεγάλη ουσία, γιατί θέλει να προστατεύσει τους Ευρωπαίους πολίτες και όσους ζουν στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης από ανθρώπους που θέλουν να εισέλθουν σε αυτήν παράνομα. Επίση, θα μα βοηθήσει στην καταπολέμηση τη απάτη που σχετίζεται με τα οχήματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να υπάρχει μια τέτοια βάση δεδομένων, να αξιοποιείται σωστά από όλα τα κράτη-μέλη και τα κράτη-μέλη να εξασφαλίσουν ότι θα προστατεύεται η ασφάλεια όλων των πολιτών και στο μέλλον. Ο κύριος Ζάκη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι. Η πλαστογράφηση εγγράφων είναι πολύ συχνά το πρώτο στάδιο στο οποίο προβαίνει κανείς ε, όταν θέλει να επιδοθεί σε ενέργειες, σε πράξεις ε, του οργανωμένου εγκλήματος. Όπως για παράδειγμα το ξέπλυμα χρήματος ή άλλες μορφές ε, εγκλημάτων τύπου μαφίας. Γι' αυτό και είναι εξαιρετικό βήμα να εναρμονίσουμε τις προσπάθειές μας όσον αφορά την καταπολέμηση αυτών των παράνομων πρακτικών και θα πρέπει πραγματικά να είμαστε πανευτυχείς που δημιουργείται αυτό το σύστημα. Εγώ δε είμαι εξαιρετικά ευτυχής που ανατέθηκε η χρήση αυτού του συστήματος στον Frontex, ο οποίος είναι ένας οργανισμός με μεγάλη εμπειρία όσον αφορά τη διαφύλαξη της ασφάλειας στην Ευρώπη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, εισηγήτρια για την εξαιρετικά σκληρή δουλειά που έκανε σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ ο Σόκολ. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Αντιπρόεδρε. Το ζήτημα της ασφάλειας είναι ένα από τα σημαντικότερα για τους ε, Ευρωπαίους πολίτες, γιατί γνωρίζουμε όλοι ότι υπάρχουν γύρω μας μια σειρά από απειλές, τρομοκρατία, οργανωμένο έγκλημα κτλ. Από αυτή την άποψη τα πλαστά έγγραφα αποτελούν μεγάλη πηγή κινδύνων, διότι δίνει τη δυνατότητα ένα πλαστό έγγραφο σε ανθρώπου εγκληματίε να εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να διαπράττουν ε, αξιόπινε πράξει ή ακόμη και τρομοκρατικέ επιθέσει. Το σύστημα λοιπόν είναι εξαιρετικό, επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών, υπάρχουν ε, εντός του συστήματος αυτού διάφορα παραδείγματα πλαστοποιημένων, πλαστογραφημένων εγγράφων και αυτό ακριβώς είναι η σωστή απάντηση όσον αφορά το ζήτημα της ενίσχυσης ασφάλειας των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ενισχυθεί ο χώρος Σέγγεν, η ασφάλεια στον χώρο Σέγγεν μέσω του συστήματος αυτού. Θέλω να ευχαριστήσω και ε, την εισηγήτρια και καλώ όλους τους συναδέλφους να υποστηρίξουν το κείμενο αυτό. κυρία Γκλάβακ, σας ευχαριστώ. Συγχαρητήρια κύριε Μητσολά για τα όσα κάνατε. Εξαιρετικό το έργο σας. Και εγώ θέλω να προσθέσω ότι το 2019 είχαμε 14.000 πρόσωπα που πέρασαν τα σύνορα ε, στον διάβλο των Βαλκανίων. Το 2018 18 η φυλακή επισήμανε πολλά έγγραφα παραποιημένα στα σύνορα. 40% περισσότερο από το παρελθόν και τα περισσότερα από αυτά τα έγγραφα είχαν παραποιηθεί, πλαστογραφηθεί με τρόπους περίπλοκους ε, και η καταπολέμηση αυτού του φαινομένου σημαίνει ότι θα πρέπει να επιστατεύσουμε ό,τι μέσα έχουμε να καταβάλουμε ό,τι προσπάθεια υπάρχει συνδυασμένη ε, συνεργασία των κρατών μελών. Και εν κατακλείδη πρέπει να σας πω ότι μία από τις προτεραιότητες της ε, Προεδρίας μας είναι η ασφάλεια. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν τέτοιες απειλές για την ασφάλεια. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Ολοκληρώνεται έτσι ο κατάλογος των αγορητών και έχουμε τώρα τη διαδικασία Catch the Eye. Έχουμε μείνει πίσω σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα, οπότε δεν θα μπορέσω να δώσω το λόγο σε όλους ε, όσοι τον ζήτησαν. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να φροντίσουμε όλοι, ε, όλες οι πολιτικές ομάδες να τοποθετηθούν μέσω των όσων ζήτησαν το λόγο. Ένα λεπτό έχει η κυρία Γραπίνη. Σας ευχαριστώ πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Όντως, το θέμα είναι πολύ σημαντικό και είναι πολύ ευχάριστο το ότι έχουμε για το φάντο αυτή την έκθεση. Ποιοι όμως είναι οι πλαστογράφοι. Δεν είναι κανένας με αγαθές προθέσεις. Πρόκειται για κάποιον ο οποίος ευθύς εξ αρχής έχει σκοπό να διαπράξει κάποιο έγκλημα. Έγκλημα, τρομοκρατία, ε, κάποιο είδους τέτοια παρανομή πράξη και οπότε θα πρέπει